Σας θερμοπαρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε, καθίστε παρακαλώ στις θέσεις σας. Συνεχίζουμε, επαναλαμβάνουμε τις εργασίες της Συνόδου. Παρακαλώ θερμά καθίστε στις θέσεις σας. Σε ένα λεπτό θα αρχίσουμε, γι' αυτό παρακαλώ καθίστε. Συνεχίζουμε τις εργασίες που είχαμε διακόψει στις 8 ε, ε, Φεβρουαρίου. Θα ήθελα καταρχήν ε, να καλωσορίσω τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Χέρμαν Βαρόπο, για πρώτη φορά στην παρθενική του εμφάνιση στην Ολομέλεια. Καλώς ήρθατε κύριε πρόεδρε. Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να προθερμαθούμε και να ξεκινήσουμε στη συζήτηση. Κανένα 15 λεπτό για τα δικαστικά. Θα ήθελα επίση να καλωσορίσω θερμά και τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Μπαρόζο, που είναι συνήθι γνώριμο στι τελευταίε ε, πενταετία. Δεν είναι καινούρια λοιπόν η παρουσία του κύριου Μπαρόζο στην ολομέλειά μα. Και θα ήθελα στην αρχή να κάνω ορισμένε παρατηρήσει, αγαπητοί συνάδελφοι. Με θλίψη καταρχήν θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι στο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έλαβε χώρα κοντά στις Βρυξέλλες έχασε τη ζωή της και η κυρία Κλάουδια Καντεάγκο, συνάδελφος από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας. Η κυρία Καντεάγκο εργαζόταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το Δεκέμβριο του 2008. Θα διαβιβάσω εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα συλληπιτήρια και τη συμπαράσταση προς την οικογένειά της. Μια άλλη τραγωδία των περασμένων ημερών ήταν οι πλημμύρες στο πορτογαλικό νησί της Μαδέρας. Η χειρότερη θεομηνία από το 1993 που κόσε τη ζωή τουλάχιστον σε 38 άτομα. Σε αυτές τις θλιβερές λοιπόν ημέρες βρισκόμαστε με τις σκέψεις και τις προσευχές μας στον πλευρό των οικογενειών των θυμάτων των δύο αυτοκαταστροφών. Θα ήθελα τώρα να σηκωθούμε και να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των δύο τραγωδιών. Dziękuję Państwu. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω εγκάρδια τους παρόντες στην αίθουσα της Ολομέλειας, τους καλεσμένους μας από τη Λευκορωσία, την κυρία Αγγέλικα Βόρης, πρόεδρο του Συλλόγου Πολωνών της Λευκορωσίας, καθώς και τον κύριο Αλέξανδρο Μιλινκέβιτς, ηγέτη της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης και βραβευθέντα με το βραβείο Ζαχάροφ το 2006. Ο κύριος Μιλινκέβιτς είναι ηγέτης Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης στην Λευκορωσία και έχει βραβευθεί με το δικό μας βραβείο Ζαχάροφ. Δυστυχώ, ε, η Λευκορωσία ξαναβρέθηκε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων εξαιτία τη δίωξη που ασκήθηκε σε μη κυβερνητικέ οργανώσει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προασπίζει ανέκαθεν τι οικουμενικέ αξίε τις ε, οποίε ασπάζεται και θα στυλιτεύει τα αυταρχικά καθεστώτα που χρησιμοποιούν την ισχύ του και τη βία και καταδιώκουν δημοκρατικέ οργανώσει μόνο και μόνο επειδή δεν εστερνίζονται τι απόψει του καθεστώτο. Σα έχουν μοιραστεί τα πρακτικά της 11 μέχρι την 11η Φεβρουαρίου. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Όχι, οπότε εγκρίνονται τα πρακτικά. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι η γραπτή δήλωση 54 του 2009 για τη μεταφορά των αλόγων για σφαγή της κυρίας Ελίζα Μεθλίν και του κύριου Κάρλ Σλούτερ της, της Συντονίας Τζεγεύσκα υπογράφηκε το 24, 24 Φεβρουαρίου του 2010 οπότε με βάση το άρθρο 123 παράγραφος 4 του κανονισμού θα διαβιβαστεί